Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το θέμα μας. Δηλαδή, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, θα ακούσουμε τον πρόεδρο Μπαρζάνη που θα μας εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση στο Κουρδιστάν, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η σταθερότερη περιοχή του Ιράκ. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τη στρατηγική που ακολουθείται για την πολιτική οργάνωση στο Κουρδιστάν. Η σταθερότητα του Κουρδιστάν είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο στη δημοκρατική ζωή του Ιράκ ολόκληρο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα ως προς τις ενεργειακές προμήθειες. Όπως θα ξέρετε, η στρατηγική της Ένωσης στοχεύει στη διαφοροποίηση των πηγών της και χρειάζεται μάλιστα σταθερές προμήθειες. Το Κουρδιστάν είναι αυτόνομη περιοχή, αυτόνομη περιφέρεια του Ιράκ, αλλά η αυτονομία αυτή πρέπει να εμφαίνεται και σε κάποιο κείμενο. Ας πούμε στη, στο καταστατικό της ε, Ομοσπονδιακής Οργάνωσης του Ιράκ. Θα τα πει βέβαια και ο κύριος Μπαρζάνη όλα αυτά. Η σταθερότητα του Κουρδιστάν λοιπόν είπα είναι κάτι το ουσιώδες για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι κουρδικοί πληθυσμοί όπως την Τουρκία και την Περσία να επωφεληθούν. Τέλος, δηλώνουμε την ικανοποίησή μας ε, για το γεγονός ότι το Ιρακινό Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποβάλει ο σχέδιο νόμου για την αλλαγή του εκλογικού νόμου που ελπίζουμε να λάβει χώρα σε πλαίσια τάξης και ηρεμίας και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους, άνδρες και γυναίκες, να συμμετάσχουν στην δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ εκ νέου τον πρόεδρο Μπαζάνη για την παρουσία του και του δίδω ευχαρίστω στο λόγο.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 Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ σήμερα. Είναι η προηγούμενη ομιλία. Και θα ήθελα να σα εξηγήσω την κατάσταση που, που επικρατεί στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτό έχει πει. Επαναλαμβάνω. Την παρουσία μου εδώ την θεωρώ μια ευκαιρία να σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα στο Ιρακινό Κουρδιστάν θα γνωρίζετε μάλλον ότι τον περασμένο Ιούλιο έγιναν βουλευτικές εκλογές. Και όλοι οι παρατηρητές, πολλοί εκ των οποίων ήταν από τις ευρωπαϊκές χώρες, άλλη ιδέα από διεθνείς μήκη όμικρον επιβεβαίωσαν ότι οι εκλογές αυτές δεν είχαν ούτε βία ούτε νοθεία. Είμαστε πολύ περήφανοι για το επίπεδο δημοκρατικότητας και εφταξίας που επέδειξε ο λαός μας κατά τις εκλογές αυτές. Συμμετέσχουν πολλές πολιτικές ομάδες και οργανώσεις, λέει ο μιλητής, καθώς και κόμματα. Πολλά της αντιπολίτευσης και με στόχο όλα να διευκολύνουν τη λειτουργία της χώρας. Έχουμε στο, στη Βουλή Κούρδους, Αρμένιδες, ε, Τουρκμένους και άλλους και όλες αυτές οι ομάδες θρησκευτικά είναι μουσουλμανικές αλλά και χριστιανικές. Τώρα αντί να σας μιλήσω για το παρελθόν και τις συμφορές του, θα προτιμούσα να πάρουμε μαθήματα από αυτό για να μιλήσουμε για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε θεσμούς στην περιοχή μας και θα ήθελα να ζητήσω και τη δική σας βοήθεια γιατί δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα πράγματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό ζητούμε τη βοήθειά σας για να υπάρξει μια επιτυχής και διαφανής διοίκηση και διακυβέρνηση ένα ευπρεπές ε, εκπαιδευτικό σύστημα ώστε τα παιδιά μας να μορφωθούν εκεί και να γίνουν ε, χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία. Καθώς και ένα υγειονομικό σύστημα, ένα σύστημα περίθαλψης. Δυστυχώς συχνά χάνονται ζωές στο Κουρδιστάν απλώς και μόνο λόγω της έλλειψης βασικών υγειονομικών αναγκών και εγκαταστάσεων και προμηθειών. Θα θέλαμε το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης στο Κουρδιστάν να αυξηθεί. Δεν λέμε βέβαια ότι θα φτάσουμε στα ίδια επίπεδα με τους Ευρωπαίους, αλλά όσο πιο πολύ, όσο κοντύτερα γίνεται. Και νομίζω ότι εσείς με τη γνώση που διαθέτετε και τα τεχνικά σας μέσα μπορείτε και σε αυτό να μας βοηθήσετε. Εκτός αυτού ζητούμε επίσης τη βοήθειά σας για να λειτουργήσει σωστότερα το δικαστικό σύστημα 30% των βουλευτών μας είναι γυναίκες. Βέβαια, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά γίνεται αγώνας και προσπάθεια στο Κουρδιστάν για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Επίσης ζητούμε τη βοήθειά σας και για την καλύτερη διακυβέρνηση γενικότερα. Όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Κουρδιστάν. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, άλλο θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η τρομοκρατία. Δεν έχει ακόμα εκκριζωθεί τελείως στο Ιράκ. Υπάρχουν ακόμη τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά τις οποίες χάνουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι. Έχουμε πάντως τη θέληση να ζητήσουμε συνεργασία και με τις ομοσπονδιακές αρχές του Ιράκ να τις βοηθήσουμε για να εκριζώσουν την τρομοκρατία. Βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει πουθενά απόλυτη ασφάλεια αλλά στο Κουρδιστάν είμαι σε θέση να δηλώσω ότι υπάρχει ικανοποιητικό βαθμός ασφάλειας και αυτό φυσικά είναι ένα ατού για την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των υποδομών. Αυτό ίσως οφείλεται τις πολιτιστικές αξίες του λαού μας που, μεταξύ των οποίων και η ανεκτικότητα. Επίσης, ο κόσμος γενικότερα στηρίζει τις αρχές ασφαλείας όποτε πρέπει να δράσουν για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Η Βαγδάτη που είναι η πρωτεύουσα του Ομοσπονδιακού κράτους είναι και δική μας πρωτεύουσα και παρά τα προβλήματα που έχουμε με την κεντρική κυβέρνηση νομίζουμε ότι το Σύνταγμα μπορεί να λύσει τις διαφορές αυτές το θέμα των ενεργειακών πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ισοκυρκούκ και πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι Πολλοί θεωρούν ότι η ολοκληρωτική ιδεολογία παραμένει ακόμη στα πνεύματα πολλών γιατί η δικτατορική διακυβέρνηση του Ιράκ ήταν καταστροφική για όλους. Το Ιράκ είναι πολύ πλούσια χώρα και νομίζουμε ότι μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό διεθνή ρόλο με ηγετική συμμετοχή σε αυτόν και του Κουρδιστάν. θα θέλαμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έρθουν και να επενδύσουν στο Κουρδιστάν γιατί μπορεί το Κουρδιστάν να αποτελέσει μια βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη ολόκληρου του Ιράκ. Ιράκ το οποίο έχει μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη και επενδύσεις αλλά μειώνονται αυτές λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί. Στο Κουρδιστάν όμως ειδικά είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τις επενδύσεις και έτσι μπορέσει, μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Τον Ιανουάριο στις γενικές βουλευτικές εκλογές νομίζω θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης του Ιράκ αλλά δεν μπορώ να προδικάσω ποιες αλλαγές θα είναι αυτές. Δεν πιστεύω όμως ότι οι διαφορές που υπάρχουν ακόμη μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και Κουρδιστάν θα λυθούν από τις εκλογές, μέχρι τις εκλογές εκείνες. Δεν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις τέτοιες μέχρι τις εκλογές. Όσο για τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες, ανέκαθεν είχαμε ως πολιτική τον αμοιβαίο σεβασμό χωρίς παρεμβατικότητες. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι έχουμε φιλικές σχέσεις με την Τουρκία και το θέμα και το ότι η τουρκική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ανοίγεται κάπως περισσότερο προς το κουρδικό θέμα είναι κάτι που μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα. Για άλλα πολιτικά θέματα οι σχέσεις μας με την Τουρκία συνεχώς βελτιώνονται και νομίζουμε ότι και αυτό θα έχει θετική επίπτωση στην γενικότερη ασφάλεια της περιοχής. θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορέσουν να επενδύσουν στο Κουρδιστάν και σας καλώ όλους να έρθετε να μας επισκεφθείτε στο Κουρδιστάν για να δείτε τα πράγματα με τα ίδια σας τα μάτια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε και ελπίζω να σας δούμε στο Κουρδιστάν. Ευχαριστώ. Καλώς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρέμβασή σας και τις απόψεις που αναφέρατε για την κατάσταση όχι μόνο στο Κουρδιστάν αλλά στο Ιράκ και τις γειτονικέ χώρες και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τη βελτίωση των σχέσεών σας με την Τουρκία σε σχέση με το Κουρδικό, κάτι το οποίο δίδει πολλές ελπίδες όχι μόνο για την περιοχή σας, για το Κουρδιστάν, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα τώρα να δώσω δυνατότητα στους συναδελφούς να ομιλήσουν, πρώτα απ' όλα στον κύριο Στίβενσον, τον πρόεδρο της Επιτροπής για τη σχέση με το Ιράκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο αυτή τη στιγμή, διότι όντως πρέπει να φύγω για να προεδρεύσω σε λίγο την αντιπροσωπεία για το Ιράκ. Αλλά θα ήθελα να χαιρετήσω τον πρόεδρο Μπαρζάνη και να του πω ότι πόσο χαίρομαι που έχω την τιμή να ε, τον ακούω σήμερα στις Βρυξέλλες συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε σχετικά με την ανάγκη για μία συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Κορδιστάν για να προωθήσουν την παιδεία, το δικαστικό σύστημα και όντως πιστεύω ότι προσβλέπουμε όλοι σε αυτή τη συνεργασία. Θα ήθελα κάτι να πω σχετικά με την επερχόμενη εκλογή η οποία προβλέπεται να οργανωθεί τον Ιανουάριο στο Ιράκ και είναι πολύ σημαντικές διότι οι πρόσφατες βομβιστικές ενέργειες το περασμένο Σαββατοκύριακο που σκότωσαν ε, ε, και τραυμάτισαν ε, πολλούς δείχνει ότι υπάρχουν συμμαχίες για να καταπολεμήσουν τις εκλογές και γι' αυτό χρειάζεται η δημοκρατική διεργασία πρέπει όλοι να καταδικάσουμε και να κηρύξουμε ε, παράνομες ε, ενέργειες αυτού του είδους. Αλλά για μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βασικό θέμα είναι μια τέτοια παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ δηλαδή από χώρες γειτονικές ε, στο Ιράκ τρίτες χώρες. Δηλαδή, κανείς δεν θα ήθελε το Ιράν να επηρεάσει πάρα πολύ τις υποθέσεις ε, του Ιράκ και μία από τις κόκκινες γραμμές ε, βέβαια είναι η παραγωγή των ε, πυρηνικών όπλων στο Ιράν, στο οποίο θα τελείως αλλά την τελευταία φορά που έγιναν εκλογές 1,5 ε, εκατομμύριο πρόσφυγες από το Ιράκ ζούσαν σε χώρες εκτός του Ιράκ και υπήρχαν ε, μόνο τρία εκλογικά κέντρα τα οποία ήταν ανοιχτά στην ε, Μέση Ανατολή, στην Ιορδανία, στη Συρία και στο Λίβανο. Υπήρχαν πάρα πολλοί πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν στην περιοχή σας 600.000 ε, πρόσφυγες και θα παρακαλούσα να προσπαθήσετε ε, όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινών προσφύγων σε Οδική Αραβία και αλλού να τους δώσετε τη δυνατότητα να εκφράσουν την ψήφο τους και αντιλαμβάνομαι ότι μόνο έξι θέσεις στο Κοινοβούλιο είχαν προβλεφθεί για τους ε, Ιρακινούς του εξωτερικού ε, ενώ υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες οι οποίοι θα γυρίσουν στη χώρα τους όταν ε, ησυχάσει η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία λαϊκή δημοκρατική κυβέρνηση η οποία θα προασπίζει τα συμφέροντα του Ιράκ και όχι κομματικά και πιστεύω κύριε Μπαρζάνη ότι είσαστε σε θέση να να παίξετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσετε ένα δημοκρατικό μέλο για το Ιράκ και να δώσετε ε, τη δυνατότητα να ψηφίσουν ε, αυτοί ε, οι Ιρακινοί του εξωτερικού. Οπότε σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας εκ προημίου. La parola a questo punto al το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Κελάν. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπαρζάνη, είμαι πολύ ευτυχής να σας καλωσορίζω εδώ και είναι μια πολύ ευχάριστη δυνατότητα που μας επιτρέπει να χαιρετήσουμε ό,τι έχετε κάνει για να σταθεροποιήσετε το Ιράκ και για να προωθήσετε τα συμφέροντα του έθνου σας όντας ένας από τους ιδιωτές του μετόπου του Κουρδιστάν και ε, έχοντας συμπράξει στις συμφωνίες του Ουάσιγκτον. Θέλω να αναφερθώ στη συνεργασία με τις διάφορες εθνότητες, διότι πέρυσι όταν ε, επισκέφθηκα το Βόρειο Ιράκ και το Κυρκούκ και το Αρμπίλ μας επισκέφθηκαν ε, διάφοροι Ιρακινοί, Χριστιανοί και Σύριοι. Ε, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ε, για καταπιέσεις, ε, για εκδιώξεις των χριστιανών από τα χωριά τους, ε, σκοτωμούς και για βέβαιο μέλλον. Επίσης, ζήτησαν να έχουν κάποια αυτονομία σαν χριστιανοί διότι είναι μία από τις πιο παλιές χριστιανικές κοινότητες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε, τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε τα συμφέροντα αυτών των μειονοτήτων. Και δεύτερον, μήπως ε, μπορείτε να σχολιάσετε την νομοθεσία για το πετρέλαιο και το αέριο, διότι υπάρχουν ακόμη ε, διαφορές, αντιλαμβάνομαι και τι σκοπεύετε να κάνετε για να τις επιλύσετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες τώρα. Thank you. Mr. President and... Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ε, Πρόεδρο Μπαρζάνη θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με όσους ε, σας επένεσαν και ε, επένεσαν και το ρόλο που έπαιξε η περιφερειακή σας κυβέρνηση ε, στην σταθεροποίηση στην περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι ε, γι' αυτό το λόγο και η έκθεση υπερψηφίστηκε εις ε, το Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που αναφέρεστε στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ιράκ και της περιοχής σας ιδιαίτερα. Μπορώ η ίδια να πω πόσο, πόσο διαπιστώσαμε ότι υπάρχει όντως μία περιοχή ασφαλής στο Ιράκ ιδιαίτερη. Θα ήθελα να σχολιάσω και τα σχόλια του κυρίου Στίβενσον σχετικά με τις ε, θετικές εξελίξεις της ε, ε, σχέσεώς σας με την Τουρκία και αντιλαμβάνουμε τώρα ότι οι τουρκικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν στο Ιράκ και ιδίως στο Καρατζίν και επίσης θα ήθελα να ακολουθήσω το σκεπτικό του κυρίου Κέλαμ, δηλαδή ε, την νομοθεσία για το πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, πράγμα όμως το οποίο δεν εμποδίζει ε, να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές σας ε, και ε, τα τάσματα αερίου. Θα ήθελα λοιπόν να τα σχολιάσετε. Συμφωνώ σχετικά με την με την κατάσταση εις το Ιράκ και ιδίως στην περιοχή σας. Ήθελα όμως να αναφερθώ και στην κατάσταση των γυναικών, διότι το 2008 όταν ε, επισκέφθηκα το κοινοβούλιο σας, μία από τις πρώτες ερωτήσεις το, τις οποίες μου έθεσαν οι εκπρόσωποι του KRG είναι, ε, ήταν σχετικά με την κατάσταση των γυναικών, διότι υπάρχουν ε, πολλές αυτοκτονίες και αντιλαμβάνομαι ότι πολύ σωστά οι εκπρόσωποι του KRG ε, εξέφρασαν αυτές τις ανησυχίες και ελπίζω ότι έχουν υιοθετηθεί μέτρα για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και τέλος θα ήθελα να σας συγχαρώ για το ρόλο που έχει διαδραματίσει και η ΑΝΤΖΗ ε, και σχετικά με τις γυναίκες ε, στην οργάνωση των ε, εκλογών και θα ήθελα να ξέρω τι θέση είχε το Κυρκούκ σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Το, το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος για να απαντήσει στον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτο το ερώτημα του αγαπητού μου φίλου Στίβενσον. Εμείς είμαστε κατά οποιασδήποτε παρέμβασης από οποιαδήποτε γειτονική χώρα στα εσωτερικά του Ιράκ. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζουμε τη δημιουργία φιλικών δεσμών με τις χώρες αυτές με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την εξυπηρέτηση αμοιβαίων συμφερόντων. Τα προβλήματα του Ιράκ πολλές φορές οφείλονται σε παρέμβαση των γειτόνων του. Γι' αυτό είμαστε κατά τέτοιων παρεμβάσεων. Όσο για την αύξηση των εκλογικών κέντρων, η Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε όποτε ζουν 20.000 ρακινή να έχει εκεί και ένα εκλογικό κέντρο. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί είναι δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Τώρα το ερώτημα του κυρίου Κίλων. τα εγκλήματα κατά των χριστιανών αδελφών μας είναι κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα και το οποίο καταδικάζουμε. Δεν πιστεύω ότι οφείλονταν στη θρησκεία τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Μοσούλη είχαν δολοφονηθεί 15 χριστιανοί από τρομοκράτες. Ταυτόχρονα 2.000 πέντε μουσουλμάνοι Κούρδοι δολοφονήθηκαν από τους ίδιους τρομοκράτες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους χριστιανούς και από τη Μοσούλη και από το υπόλοιπο Ιράκ και μέχρι 6.000 χριστιανικές οικογένειες κατέφυγαν στο Κουρδιστάν και τους δώσαμε ό,τι χρειάζονταν. 24.000 αραβικές επίσης οικογένειες κατέφυγαν στο Κουρδιστάν, χριστιανικές μάλλον, επίσης. Πολλοί επαγγελματίες, ιατροί κλπ. Χριστιανοί έχουν φύγει από το υπόλοιπο Ιράκ και πήγαν στο Κουρδιστάν να καταφύγουν. Αλλά επαναλαμβάνω δεν δολοφονούνται επειδή είναι χριστιανοί. Όλοι οι Ιρακινοί υφίστανται την τρομοκρατία. Μερικοί σκοτώνουν ως αυτό σκοπό κάνουν τις δολοφονίες, χωρίς άλλους λόγους. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τους χριστιανούς αδελφούς μας και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία στο Ιράκ και θα τους χορηγήσουμε ό,τι βοήθεια χρειάζονται. Τώρα για το πετρέλαιο και το αέριο. Θα ήθελα να εξηγήσω κάτι. Υπάρχει τον ο για το πετρέλαιο και το αέριο και υπάρχει το θέμα των εισοδημάτων που προκύπτουν από αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του Κουρδιστάν που δίνει, αντιπροσωπεύει το 17% του εθνικού προϋπολογισμού και εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει αυτό να ελέγχεται η δαπάνηση των χρημάτων αυτών, δηλαδή από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βαγδάτη γιατί έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο. Τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν από εμά για το πετρέλαιο και το αέριο δεν είναι κατά της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ διότι το πετρέλαιο και το αέριο και του Κουρδιστάν θεωρούμε ότι είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή ολόκληρου του Ιρακινού λαού. Απλά πρέπει να υπάρχει δίκαια κατανομή. Όσο για το Ζάχοφ όπου ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα τελευταία, μπορέσαμε να εξαγάγουμε 100.000 βαρύλια την ημέρα από εκεί. Και θεωρούμε ότι πρέπει να συνδεθεί το κοίτασμα αυτό μέσω του πετρελαιαγωγού που καταλήγει στο Τζιχάν και τα έσοδα να μοιραστούν από όλους τους, σε όλους τους Ιρακίνους, να υποφεληθεί και η κεντρική κυβέρνηση δηλαδή. 8 εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιήθηκαν για εξαγωγές από το Ιράκ, αλλά δυστυχώς τελικά μειώθηκε η παραγωγή. Μέχρι το 2011, εκτός από τις 100.000 βαρέλια που σας ανέφερα προηγουμένως, θα είμαστε σε θέση να παράγουμε ε, ένα εκατομμύριο βαρέλια για εξαγωγή. Και αυτό θα ωφελήσει ολόκληρο τον Ιρακινό λαό. Εμείς βοηθάμε όλους τους Ιρακινούς δηλαδή με τη σωστή πολιτική, αλλά η κεντρική κυβέρνηση στο Ιράκ δεν φέρεται δίκαια. Εμείς δεν παραβιάσαμε ούτε το Σύνταγμα ούτε τους νόμους. Αν διορθωθεί νομικά η κατάσταση αυτή, αποδεχτεί δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει κάνει λάθος, θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Ίσως αυτό απαντάει και στο ερώτημα της κυρίας Γκομές για το πετρέλαιο και το αέριο. θα συνεχίσουμε την πολιτική αυτή και για το πετρέλαιο και αέριο, είτε περάσει ο νομοσχέδιο είτε όχι, γιατί είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και είμαστε αποφασισμένοι η πλουτοπαραγωγική αυτή πηγή να ωφελήσει ολόκληρο τον Ιρακινό λαό. Δεν θα περιμένουμε όμως μέχρι να αποφασίσει η κεντρική κυβέρνηση ποια πολιτική θα ακολουθηθεί, γιατί μέχρι τώρα η πολιτική της ήταν αποτυχημένη. Ο πετρελαγωγός Ναβουχοδονόσορ έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει το Ιράκ μέσω της σύνδεσης του με το τουρκικό σύστημα. Έτσι θα μπορέσει το Κουρδιστάν να παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο, γιατί όλοι οι πετρελαγωγοί περνούν από το Κουρδιστάν, που έχει βέβαια πολλούς πόρους και κοιτάσματα, και αυτό ενδιαφέρει και την Ευρώπη όσο και μας. Όσο για τις μειονότητες στο Ιρακινό Κουρδιστάν, συμμετέχουν και αυτές στην Βουλή του Κουρδιστάν με πλήρη και ίσα δικαιώματα και όπως είπα και πριν σας καλώ να έρθετε να τα δείτε όλα αυτά να δείτε όλες τις θρησκευτικέ κοινότητες, τις μειονότητες, να συναντηθείτε ελεύθερα μαζί τους και να συνομιλήσετε και μάλιστα θα μας βοηθούσατε αν βρίσκατε καμία έλλειψη στην πολιτική μας για να τη διορθώσουμε. Όσο για τα εγκλήματα τιμής, ε, είναι λυπηρό και αυτό. Ε, στη Μέση Ανατολή ζούμε και στη Μέση Ανατολή υπάρχουν τέτοια ήθη. Η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν και η Κουρδική Βουλή έχει προσπαθήσει να απαλείψει τέτοιου είδους συνήθειες γιατί οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Έχουν επιτευχθεί πολλά αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα και τα νομοσχέδια που έχουν εγκριθεί ελπίζουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των επιθέσεων κατά γυναικών. Θα ασχοληθούν έξι ειδικέ υπηρεσίε με αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω δυστυχώ είναι και τμήμα των ηθών που επικρατούν γενικότερα. Θα προσπαθήσουμε πάντως να το απαλείψουμε. Ακόμα τρεις ερωτήσεις. Φλότρε, Χατζηγεωργίου και Μπέλτερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπαρζάνη για την παρουσία σας. Είπατε ότι η σχέση σας με τις α, τουρκικές αρχές βελτιώνονται και ότι θέλετε να έχετε ήρεμες, γαλήνιες και ειρηνικές σχέσεις με όλες τις γειτονικέ χώρες. Αγαστή πρόθεση την οποία χαιρετίζω. Στην γειτονία σας, η σχέση σας με την Τουρκία ήταν μεγάλο πρόβλημα για σειρά δεκαετιών. Υπάρχουν πολλοί ένοπλοι άνδρες του ΠΚΚ τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε το δημοκρατικό άνοιγμα που γίνεται στην Τουρκία εν ώψη μιας ειρηνικής και δημοκρατικής λύσεως του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία. Πιστεύω ότι ο ρόλος σας μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικός ακριβώς ε, για να υπάρξει δημοκρατική και ειρηνική λύση μακροπρόθεσμη για το κουρδικό. Ποια η άποψή σας από αυτού, που προφανώς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για όλους και ιδιαίτερα για την περιοχή σας. Ο κύριος Χατζιωργίου. Θέλω και εγώ κύριε Μπαρζανή να σας συγχαρώ για την σε ευθύνε που έχετε αναλάβει για την μεγάλη δουλειά που προσπαθείτε να φέρετε σε πέρας. Υγείστε ενό λαού με ιδιαίτερα και πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχουν πολλοί ηγέτες στον κόσμο που έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες σοβαρές καταστάσεις. Θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα στα, όχι, όσα έχει πει προηγουμένως η κυρία Φλότ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία με την Τουρκία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθον της ε, ευρύτερης ειρήνευσης στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν αναπτυχθούν οι σχέσεις σας με τους Κούρδους της Τουρκίας και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω με ποιο τρόπο εσείς διαπραγματεύεστε αυτό το ζήτημα των Κούρδων της Τουρκίας, πώς ενισχύετε την προσπάθεια που καταβάλλετε με αλφαϊότα για να αποκτήσουν αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων στην Τουρκία τα δικαιώματά τους. Ήμασταν πρόσφατα στην Τουρκία στα πλαίσια της Επιτροπής, Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου εκπρόσωποι των Κούρδων εκεί μας είπαν, υποστηρίζοντας βέβαια την προσπάθεια που ξεκίνησε η ηγεσία της Τουρκίας για κάποια λύση στο κουρδικό, αλλά ουσιαστικά μας είπαν ότι αυτή η προσπάθεια είναι ακόμα μία ταμπέλα δεν έχουν δικαίωμα στην γλώσσα σε σχολεία και πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Θέλω να κατανοήσω, αν μου επιτρέπετε, πώς εσείς παρεμβαίνετε στο να αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι τα δικαιώματα τους. Είπατε ότι τα προβλήματα του Ιράκ προέρχονται από τους γειτόνους τους. Σωστό και να μου επιτρέψετε να πω ότι όλα τα κράτη του κόσμου αν έχουν προβλήματα κυρίως από τους γειτόνους τους είναι όμως, στην περίπτωση του Ιράκ, και δεν πρέπει να το αποφεύγουμε να το λέμε, υπάρχουν προβλήματα και ένεκεν της εισβολής των ΗΠΑ. Δεν ξέρω τι δικαιολόγηση μπορεί να δώσει κάποιος για το ότι εισέβαλε για να τερματίσει το καθεστώς του Σάδαμ Χουσέιν, αλλά από εκεί και μπρος υπάρχει μια παρουσία δεκαετής, δεν ξέρω τι πλέον ωφελεί τον κουρδικό λαό, τον, Ιρακινό λαό, με εκατοντάδες νεκρούς σχεδόν κάθε εβδομάδα από εκρήξεις βομβών και, άλλου τέτοιου τύπου προβλήματα. Ακόμα και νεκρούς βέβαια από την ίδια την Αμερική και, την, και άλλες χώρες που συμμετέχουν. Και θέλω να κλείσω με το εξή ερώτημα. Είστε μια αυτόνομη περιοχή. Θέλετε να γίνετε κράτος και εάν ναι, πώς το προσπαθείτε και αν δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε. Κολέγα Μπέλντερ. Μπέλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Μπαρζάνι, είναι μεγάλη η χαρά μας που σας ε, ξαναβλέπουμε εδώ στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή μας ως μέλος αυτής της Επιτροπής έχω πολλές φορές μπορέσει να μεταβώ στην περιοχή σας και όπως είπατε και εσείς, ήδη η σώμαση είδα την πρόοδο που έχετε κάνει σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα από πλευράς ασφαλείας και μπορέσατε να με βοηθήσετε να κατανοήσω τους μεάνδρους της ε, Ιρακινής και κουρδικής ιστορίας. Κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά και χρήσιμο για μας. Με τον τεράστιο αριθμό προσφύγων, χριστιανών Αράβων κυρίως, έχετε αποδείξει ήδη ότι πολλά μπορείτε να κάνετε. Πώς θεωρείτε ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ρυθμιστεί η κατάσταση ίσως ό,τι αφορά τους ε, χριστιανούς. Υπάρχει θέμα αναγνώρισης με τα διπλώματα και τα προσόντα επαγγελματικής επάρκειας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι άνθρωποι να αλλαξοπιστούν. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο στο Κουρδιστάν. Μήπως θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια επ' αυτής της άποψης. Υπάρχουν πρόβλημα με το δελτίο ταυτότητας, αναφέρεται το θρήσκευμα σε αυτό, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα αναγνώρισης, ε, νομικής δηλαδή αναγνώρισης δικαστών, αλλά και κληρικών, ευαγγελιστών και άλλων. Με τα παιδιά όλων αυτών των χριστιανών προσφύγων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για την ε, ε, παιδεία τους, για τη γλώσσα τους. Έχουν βεβαίως δικαίωμα συμμετοχή στα κουρδικά σχολεία, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τη γλώσσα, διότι είναι αραβόφωνα αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να κάνουμε μια προσπάθεια για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Χρειάζονται περισσότερα σχολιά, χρειάζονται περισσότερα μεταφορικά μέσα για όλους αυτούς τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Επαναλαμβάνω, τα παιδιά των χριστιανών Αράβων που έχουν καταλήξει και καταλύσει στην περιοχή σας. Πολλά προβλήματα φτάνουν στα αυτιά μας, προβλήματα που αντιμετωπίζει η χριστιανική μειονότητα εκεί και ελπίζω ότι κάτι θα μπορέσει να γίνει για το εξαιρετικά οξύ αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος Μπαρζάνη. Madame Claude Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κυρία μου. Θεωρούμε ότι η Τουρκία εξετάζει τις αιτίες του κουρδικού προβλήματος και όχι απλώς αναφέρεται εις τα αποτελέσματα όπως έκανε στο παρελθόν και λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία γίνεται τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε, ε, δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα αλλά ε, νομίζω ότι υπάρχει μία σοβαρή εξέλιξη την οποία πρέπει να ενθαρρύνουμε και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μία λύση. Άπαξ και ε, ε, ε, εντοπίστε το πρόβλημα και βρείτε μία φιλική λύση δεν βλέπουμε γιατί θα χρειαστεί να υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις και ελπίζουμε ότι το ΠΚΚ θα μπορέσει να επαέρθει στην ε, κανονική ζωή και στην ε, πολιτική ε, απλώς επέμβαση. Γι' αυτό και προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, να μην υπάρχουν λόγοι επιβιώσεως των οπλισμένων ομάδων και των ενόπλων σειράξεων και προσπαθούμε όλα αυτά να γίνουν. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τα αποτελέσματα, αλλά έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε πει επανειλημμένως, αν η κυβέρνηση της Τουρκίας χρησιμοποιήσει μία φιλική λύση θα μπορέσουμε να τους στηρίξουμε. Βεβαίως υπάρχουν και αντιθέσεις πολλές εναντίον των προσπαθειών που γίνονται από την κυβέρνηση της Τουρκίας η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Συγχαίρουμε την Τουρκία που έκανε τις σωστές κινήσεις και θα τους στηρίξουμε. Ε, νομίζω ότι τους ε, στηρίζει όλος ο πληθυσμός, αν όχι ολόκληρος, μια πλειοψηφία και εάν ε, μπορέσουν και λύσουν το πρόβλημα με το Ιράν θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το κοινό. Τώρα όσον αφορά τον επόμενο την επόμενη ερώτηση. Νομίζω ότι η το προηγούμενο μου... η προηγούμενη μου απάντηση απάντησε και σε αυτό. Διότι στο παρελθόν υπήρχαν πολλές απειλές. Τώρα όμως με την Τουρκία υπάρχει μία πιο ήρεμη κατάσταση διαλόγου, κατανόησης και όπως έχω πει και το επαναλαμβάνω στηρίζουμε αυτή την πολιτική. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την πολιτική μπορούμε να μιλήσουμε με όλες τις ομάδες στο Κουρδιστάν ε, σχετικά με την πολιτική διεργασία ακόμη και αν στην αρχή πρόκειται για μία σύντομη κίνηση και ε, θα στηρίξουμε ε, όλες τις κινήσεις αυτές ε, για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αλλά η λύση εξαρτάται από την τουρκική κυβέρνηση και τους Κούρδους αδερφούς μας στην Τουρκία. Θα στηρίξουμε όμως την προσπάθεια για να επιτύχει. Όσον αφορά ε, την ε, κατάλυση του καθεστώτος Μπαθ ε, το 2003 η, η, η πτώση αυτού του καθεστώτος ήταν ε, σωστή διότι ήταν διδεκτατορική αλλά τα λάθη έγιναν μετά από την πτώση του καθεστώτος. Ε, δεν ήταν ε, η λανθασμένη κίνηση στο να καταργηθεί η το καθεστώς αυτό αλλά ο τρόπος το πρώτο λάθος ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με την οποία η απελευθερωτική δύναμη έγινε μία δύναμη κατοχής και ε, κατήργησε όλους τους μηχανισμούς τους κρατικούς που κατέρευσαν και ε, καταλήξαμε στο αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε σήμερα. Τα πρώτα λάθη ε, ήταν ε, το ψήφισμα 1483 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όσο αναφορά τους γείτονές μας, ε, δεν, ε, δεν ε, επεμβαίνουμε στις υποθέσεις των χριστιανών, οι περισσότεροι είναι καθολικοί, υπάρχουν όμως και ορθόδοξοι και δεν έχουμε ευαισθησίες ως προς τους ο διαμαρτυρόμενους ή τους καθολικούς δεν επεμβαίνουμε ορισμένες βέβαια εποχές δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε σε μία ενιαία αντιμετώπιση παρόλο που τους λέμε ότι ευχαρίστως να βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μία κατάσταση όπου θα ε, έχετε τη δικιά σας ε, ταυτότητα. Ορισμένες φορές ε, λέγουν ότι είναι Χαλδαίοι, Χαλδαίοι, σύρι Σύριοι, και ε, υπάρχουν διαφορετικές ε, χριστιανικές ε, σέκτες, διαφορετικές γλώσσες. Δεν μπορούμε εμείς να τους επιβάλλουμε μία ταυτότητα. Αυτοί πρέπει να επιλέξουν την εθνικότητά τους, την εκκλησία τους, την ταυτότητά τους, να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε προβλήματα με τις γλώσσες. Είμαστε ευαίσθητοι στις γλώσσες και γι' αυτό έχουμε και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πώς είναι δυνατόν να διατυπώσουμε ένα σύστημα με το οποίο ε, οι χριστιανοί μας αδελφοί θα είναι ικανοποιημένοι με την ε, εκπαίδευση η οποία τους προσφέρεται. Έχουμε προσπαθήσει εντός των δυνατοτήτων μου να τους ε, προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι η γλώσσα είναι πρόβλημα, δηλαδή ο καθένας μπορεί να εξασκεί τη γλώσσα του, να έχει παιδεία, να πάνε σε κουρδικά σχολεία, σε αραβικά σχολεία ή σε σχολεία στη γλώσσα τους. Υπάρχουν πολλά νέα χωριά τα οποία είχαν καταστραφεί και έχουν ανοικοδομηθεί θα ήθελα να τα επισκεφτώ διότι έχουμε από τον προϋπολογισμό χτίσει δεκάδες χωριών για τους χριστιανούς θα ήθελα να τα δείτε και αν υπάρχουν μεμονωμένα επεισόδια θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε και να τα επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λούνατσεκ, και Κάτσιν. Quindi la Την, ε, καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νόμιζα ότι οι εκλογές πρόκειται να γίνουν στις 21 Ιανουαρίου και αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να περάσει ε, η υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο και υπάρχει μια συμφωνία του Ιρκούκ. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε τι περιέχει ε, αυτό, αυτή η συμβιβαστική ε, συμφωνία. Επίσης όσον αφορά ε, τα πετρέλαια της περιοχής. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματα τότε πώς θα μπορέσει κανείς να προβεί σε μία κατανομή των εκμεταλλεύσεων των διαφόρων πετρελαιοπηγών τι θα γίνει ε, με, σχετικά με τη δημοπράτηση που προβλέπεται για το Δεκέμβριο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε, οι διαφορές αυτές με τη Βαγδάτη ενδέχεται να δυσκοχεράνουν αυτή τη δημοπράτηση. Η κυρία Δήμοτσεκ, ε, ευχαριστώ κύριε Μπαρζάνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και μας μιλήσατε και εγώ θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την εργασία την οποία έχετε κάνει στο Ιράκ διότι όπως είπατε είναι ένας ε, ε, ασφαλής φύλακας σταθερός και όπου μπορούν να ζήσουν και άλλοι Ιρακινοί. Έχετε έχετε ο ίδιος επηρεάσει την, ε, και δημιουργήσει τη σταθερότητα αυτή στην περιοχή σας και την χαιρετίζω. Έχω τρεις ε, σύντομες ερωτήσεις. Το ένα είναι το θέμα του πετρελαίου διότι αναφέρατε ε, το σημαντικό ρόλο που θα παίξει ο αγωγός Ναμπούκο παρόλο που ξέρουμε ότι δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν το Ιράν δεν είναι μέρος του συστήματος. Θα ήθελα να ξέρω εσείς πώς αξιολογείτε τις σχέσεις του Ιράκ με το Ιράν και τι πιθανότητες πιστεύετε ότι υπάρχουν για μία δημοκρατική ένωση με το Ιράν ε, για να συμβάλλουν εις ε, την ε, αλλαγές στο Ιράν. Επίσης, όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών στην περιοχή σας. Έχω σημειώσει ότι στην περιοχή σας υπάρχουν γυναίκες στο κοινοβούλιο, δηλαδή σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχουν πολλά κοινοβούλια που έχουν 30% γυναίκες. Εκτιμούμε πάρα πολύ λοιπόν αυτή την αθρώα συμμετοχή γυναικών πολιτικών στο κοινοβούλιο σας και σχετικά με την βία, τη βία στο σπίτι, ε, της τους σκοτομούς. Πάντοτε ε, υπάρχουν τα λεγόμενα πολιτιστικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν κάποια στήριξη την οποία θα ζητούσατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσετε τις ε, οργανώσεις γυναικών στην περιοχή σας και σε αυτούς οι οποίοι ε, στηρίζουν την ε, κατάργηση της βίας κατά των γυναικών. Θα θέλατε κάποια βοήθεια στα πλαίσια αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος θα ήθελα να πω το εξής ερωτήθηκαν, ε, τέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις για τις ε, χριστιανικές μειονότητες στην περιοχή σας και εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι χριστιανική. Έχουμε ρίζες ε, από την ε, ιδολολατρική την ε, αθεϊστική εποχή και υπάρχουν και μουσουλμάνοι και άλλες ε, θρησκείες εδώ, οπότε θα ήθελα να το αντιμετωπίσετε σαν ένα πιο γυναικό. Ο κύριος Λανσμπέργκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπαρζάνη, ε, χαιρετίζω τις ε, προσιλωμένες προσπάθειές σας για το Ιράκ θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, εφόσον υπάρχει τώρα η πολυμορφία εθνοτήτων στο Ιράκ, ε, γνωρίζουμε τα προβλήματα των ο Κούρδος στην Τουρκία. Ε, υπάρχει μία μειονότητα τα Κούρδων το Ιράν υπάρχουν προβλήματα έχετε εθνικά γνωρίζετε ότι υπάρχουν εθνικά προβλήματα σε άλλες περιοχές ευχαριστώ κύριο Κάτσιν ευχαριστώ πρόεδρε Είμαστε όλοι ιδιαίτερα ευτυχείς που μας επισκεφθήκατε και ακούσαμε με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε. Θέλουμε να έρχονται καλά νέα από το Ιράκ και όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κάποια σταθερότητα στο Ιράκ και ότι εσείς έχετε συνεισφέρει σε αυτό. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το Κουρδιστάν αποτελεί πλέον κομμάτι της λύσεως και όχι του προβλήματος στο Ιράκ. Συγχαρητήρια λοιπόν για όσα επιτύχατε μέχρι τώρα. Περνώ στο ερώτημά μου. Η περιοχή σας είπατε ότι είναι μια πλούσια περιοχή. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς έχει η οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή σας. Κάνετε επενδύσεις και στο εξωτερικό και γιατί το ερωτώ αυτό. Το ερωτώ γιατί θα ήθελα να γνωρίζω ποιο βαθμό ελευθερίας έχουν οι επενδυτές σας να δραστηριοποιούνται και εκτός της χώρας. Και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα, διότι το νότιο-ανατολικό κομμάτι της Τουρκίας είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένο. Χρειάζεται επενδύσεις. Πιστεύετε λοιπόν ότι εσείς μπορείτε να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο επενδύσεων στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας. Ο κύριος Ερδογάν πάντα λέγει ότι υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης στη χώρα του. Αναφέρει επίσης ότι είναι απαραίτητο οι γυναίκες στην περιοχή αυτή της Τουρκίας να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ε, παιδεία, στην εκπαίδευση και στην ανάληψη δημοσίων αξιωμάτων. Είναι θέμα εκδημοκρατισμού και εξυγχρονισμού της Τουρκίας, λέγει ο ίδιος ο Τούρκος Πρωθυπουργό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία με την Τουρκία επ' αυτού, μια ανταλλαγή ή με ένα πρόγραμμα κινητικότητας μέσω υποτροφιών, ας πούμε. Ευχαριστώ να προσθέσω ένα δικό μου προσωπικό συντομότατο ερώτημα. Γνωρίζετε κύριε Μπαρζανή πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της πολυφωνίας ε, στην δημοκρατία. Το θέμα των μέσων ενημέρωσης ε, θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει. Αν θέλετε να μας πείτε βεβαίως δύο λόγια περί αυτού. Η απάντηση πρώτα στον κύριο Μίλα. Με χαρά βλέπουμε ότι εγκρίθηκε ο εκλογικός νόμος πρόσφατα στο Ιακοινό Κοινοβούλιο. Το θέμα του Κυρκούκ είναι σημαντικό και θα θέλαμε να λυθεί το πρόβλημα γιατί η σχέση μας με την κυβέρνηση της Βαγδάτης και τις κυβερνήσεις της Βαγδάτης το πρόβλημα πάντα ήταν το Κυρκούκ. Θα θέλαμε να πάψει για... στην επόμενη γενιά να υπάρχει αυτό το ίδιο πρόβλημα πάντοτε. Διότι 80% των Ιρακινών ενέκριναν το Σύνταγμα με την ομοσπονδιακή του δομή και θέλουμε έτσι να λυθεί ομοσπονδιακά. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Απογραφή και δημοψήφισμα μετά. Τα τελευταία χρόνια υπό το καθεστώς του κόμματος Μπαθ πολλοί Κούρδοι είχαν εκδιωχθεί από το Κυρκουκ βιαίως και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια του τη χώρα και Τουρκμένοι επίσης. Και υπήρχε ένας νόμος ότι η ιδιοκτησία της γης βασιζόταν στο ότι ο ένας Κούρδος ή Τουρκμένος έπρεπε να αλλάξουν ταυτότητα και να θεωρούνται Άραβες για να έχουν το δικαίωμα αγοραπολισίας γης. Στις 19 Μαρτίου του 2003, οπότε και άρχισε ο πόλεμος, ο απελευθερωτικός πόλεμος του Ιράκ. Τέσσερις μέρες μετά η κυβέρνηση που πρόκειται πολύ σύντομα να πέσει, πάλι είχε περάσει ένα νομοσχέδιο για την ταυτότητα των Κούρδων, αρνούμενη την κουρδική ταυτότητα δηλαδή. Το Κυρκούκ είναι το πρόβλημα και ο λόγος είναι η ύπαρξη πετρελαιοκοιτασμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι το πετρέλαιο αυτό ανήκει σε ολόκληρο τον Ιρακινό λαό. Ορισμένοι βέβαια προσπάθησαν να εμποδίσουν τον εκλογικό νόμο λέγοντας ότι πρέπει να τεθούν ιδιαίτεροι όροι για το Κυρκούκ ή να αποκλείεται από τις εκλογές η περιοχή του Κυρκούκ ή να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τους Τουρκμένους και γενικά τους μη Άραβες. Εμείς είχαμε φέρει 6.000 Κούρδους. Είχαν γίνει προσπάθειες να έρθουν Κούρδοι από το Ιράν και την Τουρκία για να αλλάξει η δημοκρατική σύνθεση του πληθυσμού. Έτσι έλεγε η Ιρακινή κυβέρνηση τότε. Αλλά αυτά δεν ήταν αλήθεια. Σχεδόν 40% εκείνων που ήρθαν από αλλού επέστρεψαν. Όσοι λένε ότι έχουν έρθει μέχρι και 600.000 είναι ψέματα. Και προκαλούμε οποιονδήποτε μας κατηγορεί ότι φέρνουμε Κούρδους απ' έξω που δεν κατάγονται από το Κυρκούκ να το αποδείξει και τότε θα τους αποκλείσουμε από τους εκλογικούς καταλόγους. Δυστυχώς έχουν γίνει προσπάθειες τέτοιας υπονόμευσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τα εκλογικά μητρώα και τους εκλογικούς καταλόγους, να γίνει εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει καμία παρατυπία. Δεν είμαστε κατά. Οι προκαθορισμένες ποσοστώσεις, εκλογικές ποσοστώσεις για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού είναι κάτι απαράδεκτο. Ο τελευταίος τέτοιος νόμος βασιζόταν στα Μητρώα του 2009. Μετά τις εκλογές, αν ακουστούν παράπονα για οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα, θα εξεταστούν για να δούμε αν υπήρξε νοθεία. Οπουδήποτε στο Ιράκ. Θεωρούμε ότι το Σύνταγμα και το άρθρο 40 είναι η λύση για το πρόβλημα του Κυρκούκ. Τελικά το Κυρκούκ είναι μια Ιρακινή περιοχή όπως και η Βαγδάτη. Δεν πρέπει να το βλέπουμε αλλιώς. Αυτή η συμπεριφορά διαφορετικής μεταχείρισης του Κυρκούκ δεν είναι σωστή. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί μέσω του συντάγματος, όπως λέει το συντάγμα. Για το πετρέλαιο είχα ξαναπεί ότι ο πετρελαιαγωγός που πηγαίνει από το Ιράκ και περνάει από την Τουρκία. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με το Ιράν. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει καμία σχέση με το Ιράν. Περνάει από την περιοχή μας και πάει στην Τουρκία. Τι σχέση έχει το Ιράν. Αν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ιράν είναι, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. τα δικαιώματα των γυναικών τώρα. Οι γυναίκες βουλευτές μας θα έπρεπε να σας προσκαλέσουν για να δείτε ή να τις καλέσετε εσείς να έρθουν εδώ για να σας πούν μόνες τους τι νομοσχέδια υπάρχουν υπέρ αυτών στο Κουρδιστάν έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες για την ίση μεταχείριση των γυναικών με τους άντρες. Για τους χριστιανούς μας αδελφούς το δικαίωμα άσκησης της θρησκείας τους είναι κατοχυρωμένο. Και τονίζω ξανά πηγαίνετε να δείτε. Υπάρχουν εκεί γεζιντοί, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και σούνοι και σιήτες Χαλδαίοι, Ασσύριοι και όλοι έχουν ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους. Με μεγάλη περηφάνεια σας το λέω αυτό. Υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα στο Κουρδιστάν. Κύριε Λαντσμπέργκης, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με καμία εθνοτική ομάδα, ούτε με τους ούτε με Άραβες. Η περιοχή μας είναι από τη φύση της περιοχή ανάμιξης λαών. Υπάρχουν και πάντα υπήρχαν και Άραβες. 80% των Αράβων στις τελευταίες εκλογές, τοπικές εκλογές, ψήφισαν υπέρ του κουρδικού ψηφοδελτίου και όχι του αραβικού, ενώ υπήρχε γιατί και οι Άραβες και οι Κούρδοι υποφέρουν από την τρομοκρατία και το, οι κουρδικές αρχές τους προστάτευσαν όλους αποτελεσματικά. Η εχθρότητα δημιουργείται από σκοτεινές δυνάμεις. Είμαι σίγουρος δε ότι θα αποτύχουν. Όσο για τους τροκμένους έχουν τα δικαιώματά τους, έχουν δικά τους σχολεία, τηλεοπτικούς σταθμούς, κόμματα και βουλευτές. καθώς και Άραβες φυσικά στα τοπικά δημοτικά συμβούλια και οι περιοχές που θεωρούνται αμφιλεγόμενες θα προστατευτούν και αυτές όταν και αν αποτελέσουν επισήμως τμήμα του Κουρδιστάν. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και τη συμβίωση ειρηνικά μαζί τους. Για τα πανεπιστήμια τώρα. Τα πανεπιστήμια μας έχουν δώσει υποτροφίες σε Κούρδους στην Τουρκία, στη Συρία, από την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράν. Και πολλοί φοιτητέ έρχονται και σπουδάζουν στο Κουρδιστάν. 400 τουρκικές εταιρείες δρούν στο Κουρδιστάν από την άλλη και 5 δισεκατομμύρια δολάρια αντιπροσωπεύουν οι εμπορικές εναλλαγές με την Τουρκία. Αυτό φυσικά βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο και το εμπόριο του Κουρδιστάν και παραμεθορίως μεταξύ Κούρδων του Ιράκ και της Τουρκίας δηλαδή. Και αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ανύψωση του βιωτικού επίπεδου του Ιρακινού Κουρτιστάν. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, εκεί υπάρχει πλήρης ελευθεροτυπία. Το σχετικό νομοσχέδιο χορήγησε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τους δημοσιογράφους, τον γραπτό και τηλεοπτικό τύπο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το Υπάρχουν δεκάδες τηλεοπτικών σταθμών, εκατοντάδες ε, ε, περιοδικών και εφημερίδων και δελτίων που δημοσιεύονται χωρίς κανένα πρόβλημα λογοκρισίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε <clears throat> για την ε, ευγένεια και την σαφήνεια με την οποία απαντήσατε στα ερωτήματα των συναδέλφων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία προσωπικά και στη χώρα σας. Ευχαριστώ και πάλι. Please, Σας παρακαλώ, πρέπει να συνεχίσουμε. Όσοι έχουν καμιά άλλη δουλειά να την κάνουν εκτός εθούσης. Τώρα περνάμε στο σχέδιο έκθεσης για σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου και για το χρηματοδοτικό μέσο κτλ. για την προαγωγή της δημοκρατίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίω. Ε, έχουμε δύο εισηγητές. Την κυρία Κίνγκα Γκάλ και την κυρία Βαρβάρα Ρόχμπιλερ. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ πρώτη. Ευχαριστώ. αποφασίσαμε με, τον, με την συνάδελφο να μιλήσουμε και οι δύο και γι' αυτό ίσως να πούμε τα ίδια πράγματα δυο φορές, αλλά έτσι είναι πιο εύκολο νομίζω να καταλάβετε τι συμβαίνει με την έκθεση αυτή που άρχισε ως καθαρά τεχνική. Πρώτον λοιπόν, η διάσκεψη των Προέδρων δεν έδωσε την άδεια συνεισηγεσίας για την έκθεση αυτή και γι' αυτόν τον λόγο καθυστέρησε ο καθορισμός των εισηγητών. Γι' αυτό και δεν μπορέσαμε να την μοιράσουμε, να τη διανύμουμε νωρίτερα και να γίνουν εγκαίρως οι μεταφράσεις. Τώρα, Ποιο είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ένα από τα επτά χρηματοδοτικά εργαλεία εξωτερικών δράσεων της Ένωσης για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες. Αντίθετα όμως από άλλα ανάλογα εργαλεία δεν χρειάζεται συμμετοχή της κυβέρνησης των τρίτων αυτών χωρών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προώθη, αποτελεσματικότερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δραστηριότητα της Ένωσης για την προώθηση των μήκη όμικρων σε τρίτες χώρες. Άργησε πολύ να λειτουργήσει βέβαια και ελπίζω οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να το επιβεβαιώσουν το φθινόπωρο του 2008 άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη το εργαλείο ή μέσο αυτό και ξέρουμε απλώς ότι συμμετέχουν πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει μία τεχνική μόνο τροποποίηση που αφορά το κόστος ε, που θα προέρχεται από δασμούς και φόρους για το μέσο αυτό. Από ό,τι καταλάβαμε είναι σημαντική η τροπολογία αυτή για να μπορέσουν οι μήκοι όμικρον να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πράγματι τις δυνατότητες που περιλαμβάνει, που προβλέπει το μέσο αυτό. Και είμαστε υπέρ της τροπολογίας αυτής της ομισιών. Η έκθεσή μας βασίζεται κυρίως σε τρία είδη τροπολογιών, σε τρεις ομάδες τροπολογιών. Η πρώτη είναι τρεις τροπολογίες και στοχεύει το διαχωρισμό της διορθωτικής πρότασης της Κομισιόν κόμμα και ζητούσε να χωρίσει το μέσο σε, να βασίζεται σε δύο διαφορετικούς κανονισμούς. Γιατί το πρώτο τμήμα, το DCI που λέμε, DCI, καλυπτόταν από μια άλλη επιτροπή, την Επιτροπή ΑΝΑΠΤ, ΔΕΒΕ. Και μετά το άλλο τμήμα κάλυπτε καθεαυτό το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Προώθηση της Δημοκρατίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άλλο θέμα που είχε τεθεί ήταν ε, και είχε πολύ συζητηθεί ήταν, λέγω, ήταν ένα οριζόντιο θέμα, δηλαδή η δυνατότητα να ενισχυθεί το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό συμπεριλάβαμε στην αρχικά καθαρά τεχνική αυτή πρόταση της Κομισιόν τροπολογίες που ζητούν απαιτούν κανονιστικές διαδικασίες και ελεγκτικές για να ενισχυθεί το ρόλος και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή ΑΝΑΠΤ επίσης το ζήτησε. Και επειδή αυτό ενισχύει όπως είπα τρεις φορές το ρόλο του Κοινοβουλίου Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε και οι δύο εισηγητές, δηλαδή οι εισηγήτριες μάλλον, ότι είναι καλό. Θα συμμεθυμίζω ότι το θέμα είναι το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίω. Αλλά βέβαια και η νομική υπηρεσία πρέπει να χρηματοδοτήσει για να είμαστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το εργαλείο αυτό, το χρηματοδοτικό εργαλείο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων παγκοσμίω έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο. Πρόκειται για ένα νέο μέσο και δεν είναι ακόμη καιρός να το αξιολογήσουμε εις βάθος αλλά συμφωνούμε με την ε, πρόταση ε, να παρουσιάσουμε ε, το πλαίσιο και να το χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών. Έχουμε πολύ τεχνικό κείμενο μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία τεχνική τροποποίηση σχετικά με τις φορολογίες και τον που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αυτού του εργαλείου. Δεν έχει προβλεφθεί καμία εξαίρεση και θα ε, επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν σε εξαιρετικές συνθήκες προγράμματα. Ε, πράγμα το οποίο δεν αντιμετωπίζει ε, αντιρρήσεις ή αντιδράσεις από το Συμβούλιο και γι' αυτό χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έπρεπε να έχει εκδηλωθεί ε, ενωρίτερα και που σέβεται το δικαίωμα εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, το 2006 έχει ε, από το 2006 ε, ισχύει η εξέταση βάσει δύο κριτηρίων εφόσον δηλαδή τα μέτρα είναι γενικά και τροποποιούν μη ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού. Ε, γι' αυτό και θεωρούμε ότι ε, έτσι ενισχύεται η δύναμη του Κοινοβουλίου και ε, ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει τροποποιημένη πρόταση και τα κριτήρια αυτά βοηθούν όσον αφορά τα ειδικά μέτρα προβλέπονται, ε, προβλέπεται ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μέτρα για την εφαρμογή της διαδικασίας RPS αυτή η διαδικασία προτείνεται πολύ αργά για να μπορέσει ε, να συμβάλλει στην τριμερή διαβούλευση των υπευθύνων ε, για την θέσπιση των χρηματοοικονομικών μέτρων και ε, τώρα δίδεται η ευκαιρία ε, να ε, ευθυγραμμιστεί η επιτροπολογία με τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Δεν προβλέπεται η έκθεση αυτή να ισχύσει πριν την αρχή ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας και θα προτιμούσαμε η έκθεση αυτή να ψηφιστεί στην Επιτροπή πριν ε, την 1η Δεκεμβρίου για να ε, διακηρύξουμε τη θέση του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στη διαδικασία συναπόφασης. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Ρικάρντο Πάσος να μας παρουσιάσει εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας την άποψή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ε, εισηγήτριες. Η κανονιστική διαδικασία με υποπτία είναι με έλεγχο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι οι αλλαγές αυτές συμπληρώνουν τη βασική νομική πράξη και αφορούν μη ουσιαστικά στοιχεία αυτής. Για τα έγγραφα στρατηγικής είναι σαφές αυτό ότι ισχύει και θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει και μια ιεραρχία μεταξύ των διαφορών κειμένων. Το ίδιο το μέσο, πρώτα απ' όλα, που εγκρίνεται μέσω συναπόφασης και τα στρατηγικά από την άλλη έγγραφα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δικαίωμα βέτο εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Άρα Καταλήγοντας θα έλεγα ότι συμφωνώ πλήρως με τις εισηγήτριες και θεωρώ πολύ καλό ότι πλέον υπάρχει μια κοινή στρατηγική η κανονιστική διαδικασία για, τις περισσότερες, ε, για τα περισσότερα μέσα στο δεύτερο τις δράσεις, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη και συνεργασία έχουν εγκριθεί για τη σταθερότητα όχι ακόμα, αλλά είναι πολύ καλό λέγω που υπάρχει ομοιογενής προσέγγιση. Συμφωνώ με τις εισηγήτρες ότι αφορά τη μετάβαση προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πολύ καλή στρατηγική αυτή του Κοινοβουλίου να έχει έτοιμη την κανονιστική διαδικασία και πριν την επίσημη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, διότι όταν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη θα είσαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. Εγώ. Ωραία. Και τώρα αν δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, ο κύριος Μίλλερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ τις εισηγήτριες για την υποστήριξη τους προς την πρότασή μας και για την τεχνική τροπολογία που αφορά στους φόρους και δασμούς. Τη δεχόμαστε. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι θα διεκπαιρεωθεί σύντομα και θα εγκριθεί το κείμενο για να μπορέσουν από του χρόνου να εφαρμοστούν επιτέλους τα προγράμματα που καλύπτει. Βέβαια τώρα μόλις διαβάσαμε το σχέδιο έκθεσης, την γνωρίζαμε την τροπολογία ήδη από πριν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι η Επιτροπή σας θα ζητήσει τις ίδιες αλλαγές και αυτό θα μας θέσει ιδιαίτερα προβλήματα γιατί η Συμφωνία του 89 ως προς την Επιτροπολογία αλλάζει το. Είχε συμφωνηθεί τότε και τώρα την αλλάζεται. Παρά τη συμφωνία για την περίοδο 2007-2013 όπου, για την οποία όλα τα όργανα είχαν συμφωνήσει τέτοια σοβαρού ύψους προγράμματα να εφαρμόζονται από την διαδικασία των διαχειριστικών επιτροπών. Και το προηγούμενο, η προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου είχε εκφράσει τις ίδιες ανησυχίες, δηλαδή σε τέτοιου είδους εργαλεία και μέσα η Κομισιόν να έχει το δικαίωμα, όπως είχε ζητήσει, να εγκρίνει στρατηγικά προγράμματα και έγγραφα, ενώ τώρα επιμένεται για συναπόφαση και για τα έγγραφα σχεδιασμού και στρατηγικής. Τελικά όμως αυτό είχε ζητηθεί και είχαμε συμφωνήσει το σύστημα της επιτροπολογίας να ακολουθήσει τη διαδικασία των διαχειριστικών επιτροπών. Και επίσης είχε συμφωνηθεί για τα στρατηγικά έγγραφα να υπάρχει δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο, δηλαδή το Κοινοβούλιο να την χάνει διαβούλευσης για αυτά τα έγγραφα, να παίρνουμε υπόψη πολύ σοβαρά τις απόψεις σας σε διαβούλευση αυτή και ο, όταν εγκρίνει ψηφίσματα όπως έχει κάνει και στο παρελθόν για τέτοιου είδους στρατηγικά προγραμματικά έγγραφα τα ψηφίσματα αυτά λαμβάνονταν πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη από εμά. Γιατί είναι μάλιστα και βασικό θέμα που καλύπτουμε και στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Τώρα όμως προτείνεται σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες του εργαλείου για τις βιομηχανικές χώρες αλλαγή που βασίζεται σε αυτή την ιδέα του δημοκρατικού ελέγχου την οποία δεχόμαστε, θέλουμε το κοινοβούλιο να εκφράζεται και όπως είπα πολλές φορές παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις απόψεις του. Σημείωσα τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και εμείς θα ζητήσουμε διαβούλευση από τη δική μας νομική υπηρεσία αλλά φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα από την αλλαγή του νομικού υποβάθρου που προτείνεται και αυτό θα βλάψει όλους τους ενδιαφερόμενους γιατί όσο αργότερα εγκριθούν τα κείμενα αυτά τόσο αργότερα θα αρχίσει και η χρήση του προϋπολογισμού τους ενώ εμείς θέλουμε να εγκριθούν τα μέσα αυτά, τα εργαλεία αυτά όσο δυνατόν συντομότερα ενώ το Κοινοβούλιο τώρα βλέπω ότι ξαναρχίζει αυτή τη συζήτηση για την επιτροπολογία και το δημοκρατικό έλεγχο και άρα θα υπάρξει τεράστια καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω ότι άκουσα τα επιχειρήματα της νομικής σας υπηρεσίας, αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μέτρα γενικής εφαρμογής, και δεν τροποποιούν τους κανονισμούς που μόνο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να τροποποιήσουν. Είναι απλώς διαχειριστικά μέτρα. Αφορούν καθαρά την εφαρμογή του εργαλείου και για αυτούς τους λόγους νομίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να τα διαχειρίζονται οι αρμόδιες οι διαχειριστικές επιτροπές. Έχουμε συμφωνήσει για το δημοκρατικό έλεγχο με τη συμφωνία 7 με 13. Θα μπορούσατε να αλλάξετε εκείνη τη διαδικασία αν, αν τίποτα δεν σας αρέσει. Ξαναρχίζοντας αυτή τη συζήτηση που νομίζαμε ότι είχε λήξει για μέχρι το 2013 θα αρχίσει μια τεράστια συζήτηση και θα καθυστερήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων. Πράγμα το οποίο θα είναι αρνητικό νομίζω για τον προϋπολογισμό από του χρόνου, αν χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη ώσπου να λυθούν τα νέα αυτά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, που μας παρουσιάσετε τις απόψεις ε, της Επιτροπής και τώρα από την κυρία Κομέσου να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω το, τις ε, συνεισηγήτριές μας. Συμφωνώ με τη γραμμή που ακολουθούν. Ιδίως βάσει της γνωμοδότησης νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και βάσει της πείρας μου, διότι έχω συμμετάσχει στην εξέταση της DCI ε, στο παρελθόν. Θεωρώ ότι ευθυγραμμίζεται αυτό πλήρως με τις ε, ευθύνες που θα ανατεθούν από τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του και το βαθμό το, τον όγκο εργασίας που θα επιβάλλει αυτή η εξέταση το κοινό ε, Βούλιο είναι έτοιμο για να αναλάβει αυτή την εργασία όπως αποδεικνύει η έκθεση και χρειάζεται πολύ πιο ουσιαστικά επιχειρήματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να ακολουθήσει διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία προτείνουν οι συγγήτριες ίσως είναι ε, επιχειρήματα τα οποία βολεύουν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή απλώς διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται απλώς στο ε, χρόνο της διαδικασίας. Εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές επιφυλάξεις θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ουσιαστικές. Ε, διότι από τα στοιχεία που έχω ε, μπροστά μου τώρα δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τις συνεισηγήτριες. Ωραία. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω τις ε, δύο εισηγήτριες να δευτερολογήσουν πρώτα η κυρία Γκάλ και μετά η κυρία Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε με τα προσοχή στα σχόλια της νομικής υπηρεσίας και της εκπροσώπου της Επιτροπής και ε, θεωρώ ακόμη και ευχαριστώ την κυρία Γόμες η οποία μας στηρίζει ότι αυτή η διαδικασία την οποία ζητάμε ενισχύει πάρα πολύ τις ε, ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε σε ό,τι παρουσιάζει υπομορφή προτάσεως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν είχαμε προβλήματα με αυτό το εργαλείο το χιμιπι ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ, αλλά θεωρούμε ότι στο μέλλον μπορεί η κατάσταση να αλλάξει. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί και γι' αυτό θεωρώ ότι οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να ισχύσουν επί της ίδιας βάσεως για όλα τα εργαλεία. Και αυτό όσον αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής διαδικασίας το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό θα καθυστερήσει τη διαδικασία και θα δημιουργήσει προβλήματα και εγώ συμφωνώ ότι για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και για την κοινωνία των πολιτών που θα επωφεληθεί από αυτό το εργαλείο είναι πολύ βασικό η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υιοθετεί αλλά γιατί την ε, παρουσίασαν μόνο τώρα εφόσον το πρόβλημα έχει προκύψει από την αρχή του παρελθόντος έτους οπότε δεν νομίζω ότι ε, η καθυστέρηση οφείλεται στο Κοινοβούλιο και ούτε ότι θα επηρεάσει πολύ το όλο θέμα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι βασικό να υποφεληθούμε της ευκαιρίας, να προχωρήσουμε και να ζητήσουμε να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες για όλα τα εργαλεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν συζητήσαμε τις τροπολογίες, συζητήσαμε και την δυνητική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε ότι θα υπήρχαν προβλήματα δεν έχουμε όμως υπερβεί τόσα σοβαρά προβλήματα και δεν άκουσα κάτι το οποίο είναι δυσεπίλητο. Οπότε επαναλαμβάνω αυτό που είπε η συνάδελφός μου, ότι από πλευρά του Κοινοβουλίου είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Επιτροπή όπου μπορούμε και θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά ε, όπως ε, λέγεται σε αυτή την τροπολογία να μην υπάρξει ε, καθυστέρηση για την εφαρμογή του εργαλείου γιατί ε, είναι πολύ εύκολο να προβεί κανείς σε εξαιρέσεις. Εμείς είμαστε υπέρ των τροπολογιών και ζητούμε να βρεθεί μια λύση ή η Επιτροπή τουλάχιστον πρέπει να βρει μια λύση το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση εδώ και η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 13 Ιουνίου το 12 το μεσημέρι. 13 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Δεν έχετε δηλαδή ακόμη πολύ χρόνο. Νοεμβρίου, με συγχωρείτε. Ε, επίσης όσον αφορά την ε, πρόταση ψηφίσματος ε, για τις ε, ε, για τις βιομηχανικές χώρες ε, προτείνω στην κυρία Λόχ Μπίλερ να επανέλθει εις ε, την ε, εξέταση του χρηματοδοτικού μέσου το οποίο θα αποτελέσει ένα βασικό μηχανισμό διότι στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο όργανο για να καλύψει ένα κενό ε, αλλά ε, περιοριζόταν μόνο στην αναψυξιακή βοήθεια η οποία είναι προς όφελος των ε, εμπλεκομένων χωρών. Οι δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΑΣ και γι' αυτό προτάθηκε να ε, τροποποιηθεί το εργαλείο για τις πολύ μικρές ε, βιομηχανικές χώρες ε, όπως και το μέσο της συνεργασίας με τρίτες χώρες και έχει προταθεί μια τροποποιημένη πρόταση χωρίς όμως να προσαρμοστεί ο τίτλος και επειδή ιστορικά το εργαλείο αυτό αυτό ήταν ε, της αρμοδιότητας της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και ε, ε, είχε ε, ε, ανατεθεί σε μία επιτροπή. Το ίδιο ε, έγινε και στην ανάθεση από το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή τώρα όπου η ΑΦΕΤ, δηλαδή η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων απλούστατα θα κάνει συστάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από την ίντα. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ ε, των δύο προέδρων Αλβερτίνη και Γουερέρα ε, δεχτήκαμε την τροποποίηση της διαδικασίας αφού όμως ε, εξασφαλίσαμε ότι δύο επιτροπές θα συνεργαστούν στενά και η ΑΦΕΤ μετά την υιοθέτηση θα συμμετάσχει στην δημοκρατική στον δημοκρατικό έλεγχο. Με τα μέτρα του Δεκεμβρίου θα αλλάξει τελείως η κατάσταση και με το άρθρο 181 από ε, διαβούλευση περνάμε σε συναπόφαση και το άρθρο 181 181α ε, ε, αναφέρεται μόνο στις βιομηχανικές χώρες και δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει τη μοναδική νομική βάση. Επίσης τα περισσότερα εργαλεία διεθνών σχέσεων έχουν ε, διπλή ε, νομική βάση Δηλαδή ε, προστίθεται και το άρθρο 179 για την συνεργασία της υποανάπτυξης χώρες και ε, η συνεργασία με τις τρίτες χώρες ε, αναφέρεται ε, εδώ στην αναπτυξιακή βοήθεια ε, όπου όμως το μόνο θέμα το οποίο πραγματεύεται είναι η μείωση της φτώχειας και ε, πρέπει να συγχρόνως να προωθήσουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να εντάξουμε τις ανάπτυξη χώρες εις ε, την παγκόσμια οικονομία και τα στοιχεία αυτά έχουν διαγραφεί από το κείμενο και μετά τη Λισαβόνα δεν υπάρχει ε, κανένα στοιχείο για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες όπου θα μπορούσαμε να βασίσουμε αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί απλώς να παρεμβαίνει εις ε, την ανακούφιση από τη φτώχεια ή στην χρηματοδότηση σε ε, βιομηχανοποιημένες χώρες. Βλέπουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας παρουσιάζει σαφώς ένα κενό και δεν υπάρχει καμία νομική βάση για εξωτερικές σχέσεις στη συνθήκη. Σύμφωνα λοιπόν με την συνηθισμένη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αποσύρει την πρόταση αυτή και να μας παρουσιάσει ένα νέο κείμενο με νέα νομική βάση και αυτή είναι η θέση στην οποία είχα συμφωνήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ε, ε, κύριο Σόλτς αλλά ε, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες ε, πληροφορίες και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες διατάξεις για τις ε, κοινοτικές πολιτικές, δηλαδή την διάσταση εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικές πολιτικές όπως είναι η έρευνα, το περιβάλλον και άλλες και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το νέο εργαλείο με μία μακροπρόθεσμη προοπτική, ιδίως όσον αφορά τη νέα αρχιτεκτονική των εξωτερικών σχέσεων και των σχετικών ε, διατάξεων. Και επίσης ε, θα πρέπει ορισμένα θέματα να επιληθούν αφού υπάρξει νομική βάση. Ε, το εργαλείο το οποίο θα χρειαστεί να διατυπωθεί. Θα θέλαμε να μπορεί ε, να μην ε, μεταφερθούν πόροι από το DCI, από το ΕΑΣ e και ε, καταρχήν δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, μεταφορά ε, χρημάτων από την αναπτυξιακή βοήθεια για την κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών. Θα θέλαμε να αλλάξουμε και την επικεφαλίδα, παραδείγματο χάρη συνεργασία με τρίτες χώρες για μέτρα που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία ΕΑΣ. Και ε, αντί να υιοθετήσουμε το παλιό εργαλείο θα πρέπει να ε, παρουσια... Ε, θα έπρεπε να πούμε ότι η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της με πολύ πολύ πρόχειρο τρόπο και πρέπει ακόμη να γίνουν πολλές προσαρμογές για να μπορέσουν να προσαρμοστεί ο στόχος και προσβλέπω στη συνεργασία επί του περιεχομένου μαζί με τον εισηγητή του, της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ για να μπορέσει να υπάρξει πλήρη συνεργασία. Και τώρα ζητώ από τον κύριο Ρικάρδο Πάσος να μας παρουσιάσει τη νομική του συμβουλή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι συγγήτριες μου διευκόλυναν πολύ τα πράγματα. Η κυρία Λόχ Μπίμπλερ είναι ίσως οικηγόρος μάλιστα, γιατί ανέφερε πολλές νομικές λεπτομέρειες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε, απλώς θα σας πω τη δική μου άποψη. Το θέμα είναι ήδη λίγο μπλεγμένο, χωρίς να αναφέρουμε καν τη συνθήκη της Λισαβόνας και το άρθρο 181 όπως προτείνει η Κομισιόν για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόσφατα δήλωσε σε μια υπόθεση προσφυγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το 181 δεν αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος πάντων, το Κοινοβούλιο με βάση αυτή την απόφαση έκανε την πρότασή του. Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη από τον επόμενο μήνα, αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι η πρόταση αυτή επειδή, όπως είπαν οι συγγήτριες, αλλάζει το νομικό, τη στο διαδικασία νομικό υπόβαθρο, από την απλή διαβούλευση με το Κοινοβούλιο στη συναπόφαση, γι' αυτό η Κομισιόν μόλις αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να στείλει στο Κοινοβούλιο ολόκληρο κατάλογο ψηφισμάτων και εκθέσεων που θα πρέπει να εξεταστούν με τη νέα διαδικασία. Παραμένει το θέμα του νομικού υποβάθρου λοιπόν. Καταρχήν δεν μπορώ, είμαι σε θέση να σας πω σήμερα τώρα ποιο πρέπει να είναι το νομικό υπόβαθρο, διότι αυτό αφορά, σχετίζεται με το στόχο της κάθε πρότασης. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε την πρόταση για να ξέρουμε και αν είναι κατάλληλη η νομική βάση που έθεσε η Κομισιόν. Το βέβαιο είναι ότι το 182 της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί όπως είπε και η κυρία Λόχ Μπίμπλερ, αυτό αποκλείει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ποια να είναι λοιπόν η νομική βάση, θεωρητικά τα λέω βέβαια. Θεωρητικά. Λοιπόν, δύο δυνατότητες υπάρχουν. Η μία θα ήταν να συνεχίσουμε με την γνωστή τεχνική της Κομισιόν, δηλαδή να τροποποιείται η υπάρχουσα πρόταση εκ των υστέρων με διπλή νομική βάση 209 και 182 μαζί. Εδώ όμως το πρόβλημα είναι ότι η χρησιμοποίηση του 209 απαιτεί ερμηνεία διότι στη συνθήκη της Λισαβόνας το 209 λέει ότι ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Αν αναφέρεται ρητά ότι είναι από τους κύριους στόχους του κειμένου, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, τότε θα καλυπτόταν από το 209. Αυτή θα ήταν λοιπόν η πρώτη δυνατότητα να συνδυαστεί το 209 με το 182. Δεύτερη δυνατότητα να υπάρξουν νομικές βάσεις ανατομέα, δηλαδή να μην ακολουθήσουμε την τεχνική της Κομισιόν τροποποίησης του υπάρχοντος κανονισμού, αλλά να γίνει χωριστός κανονισμός με διάφορες τομεακές νομικές βάσεις. 165 για τον αθλητισμό, 167 για τον πολιτισμό και 186 για την έρευνα και την τεχανολογία γιατί όλα αυτά αφορούν συνεργασία με τρίτες χώρες χωρίς να αναφέρεται αν είναι αναπτυσσόμενες ή όχι. Αλλά ανατομέα, όχι αναπτυξιακό εργαλείο καθεαυτό δηλαδή, αλλά ανατομέα αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Αλλά το είπα και πριν πρόεδρε, θέλω να επιδείξω κάποια φρόνηση εδώ γιατί αυτά όλα είναι θεωρητικά πρέπει να ξέρουμε το περιεχόμενο της κάθε πρότασης. Ευχαριστώ κύριε Γκάλετ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι σαφές ότι αλλάζουν τα πράγματα με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Η εξωτερική πολιτική όμως ενδυναμώνεται με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξωτερικές δράσεις. Από τη μία, από την άλλη όμως υπάρχουν περιορισμοί επί τη βάση του άρθρου 212 το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα συγκεράσουμε αυτά, πώς θα μπορέσουμε να τα συμφιλιώσουμε. Όπως είπε ο κ. Ντάσας, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παράγραφους 208 ε, και 209. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τομεακές ε, πολιτικές και για τις τομεακές πολιτικές υπάρχουν ε, δεσμοί σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ε, πολιτικών. Αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις ε, ε περιπτώσεις. Δεν καλύπτει, ας πούμε, την αναπτύξη της υπαίθρου, τον τουρισμό ε, και... άλλα θέματα. Όλα αυτά δεν συνδέονται, δηλαδή, με την εξωτερική πολιτική. Μια τομεακή, λοιπόν, προσέγγιση επί τη βάση των υφιστάμενων κανόνων θα ήταν, νομίζω, ανεπαρκής. Εγώ θα ήθελα να είμαστε σε θέση να ασκούμε εξωτερική πολιτική και εναντί τρίτων χωρών. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω ε, την λύση των ε, παραγραφών 208 και 209. Ο κύριος Σούλτς, ο οποίος είναι ε, και εισηγητής στην ΕΙΤΑ, πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να λάβω το λόγο στην Επιτροπή αυτή. Στην Ήτρα δεν έχουμε βρει ακόμα συμφωνία για την έκθεση αυτή. Έγινε μια αλλαγή σήμερα στην ημερήσια διάταξη και θα επιστρέψω αμέσως μόλις φύγω από σας ε, στην ε, συνεργασία της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ ε, σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν θα ήθελα να πω ότι μας ενδιαφέρει πολύ η παρακολούθηση της καταστασής επί τη βάση της συστάμενης νομικής βάσης προσπαθούμε να εντοπίσουμε με μια λύση για να κατανοήσουμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της συναπόφασης τώρα που υπάρχει πια στον τομέα αυτό για να βρούμε μια συμφωνία στα πλαίσια του υφισταμένου μέσου. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως είπαν οι συνάδελφοι, η κατάσταση θα αλλάξει. Συμφωνώ με την συνεισηγήτρια, την κυρία Λόχομπιλ. Είναι όντως ε, απαραίτητο να γίνει μια πρόταση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, τη θέση του Συμβουλίου και πιστεύω, πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και το Συμβούλιο να τοποθετηθεί προς την Επιτροπή. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία που δίδεται τώρα να τοποθετηθεί σχετικά με τις θέσεις μας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στις ε, διάφορες επιτροπές και είναι παρεμφερείς άλλωστε, κατά τρόπον ώστε να επωφεληθεί Τη της ε, νέας νομικής κατάστασης και να μπορέσει να ενισχύσει τη θέση του Κοινοβουλίου σε συντονισμό με το Συμβούλιο. Ε, γι' αυτό και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και προσβλέπω στην συνεργασία με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε ε, τη θέση μας όσον αφορά ένα πολύ βασικό, μια πολύ βασική πτυχή των ε, θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εντάχει να πω ότι συμφωνώ με τις απόψεις που ανέφερε η κυρία Λόχμπιλ και επί της ουσίας και επί του τύπου. Θεωρώ ότι το μέσο των εξωτερικών σχέσεων θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εξωτερικής πολιτικής. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή εδώ η Επιτροπή να αναλάβει ε, την σχετική ευθύνη. Και το δεύτερο, ε, συμφωνώ ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια νομική βάση κατάλληλη ε, εις ό,τι αφορά την κάλυψη από αυτή την άποψη συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι θα πρέπει να προσεστεί ένα νέο κείμενο για το μέσο των εξωτερικών σχέσεων που να βασίζεται σε πιο στέρεες νομικές βάσεις και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της επί του θέματος αυτού διότι θεωρώ ότι είναι απολύτως κέρια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μίλλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαστε και πολύ τυχεροί με την ενδιάμεση έκθεση. Προβλήματα επιτροπολογίας και τώρα προβλήματα νομικής βάσης. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επί της δεν έχουμε ακόμα αποκρισταλώσει άποψη. Έχουμε επίγνωση του προβλήματος, εργαζόμεθα για να καταλήξουμε σε μια θέση και με τις άτυπες επαφές με τους δικηγόρους των διαφορών θεσμικών οργάνων. Δικηγόρους εννοώ νομομαθείς με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Πάσος και όποιες και αν είναι οι λύσεις ε, που θα προκριθούν ε, τελικά η συναπόφαση βεβαίως δεν αφισβητείται από κανέναν. Εις ό,τι αφορά τώρα το πώς ε, θα εφαρμοστεί αυτή η λύση, μία εναλλακτική είναι η Κομισιόν όντως να υποβάλει νέα τροποποιημένη πρόταση θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ο κύριος Σόλτς ανέφερε και την σημασία της συζήτηση του θέματος και με το Συμβούλιο, διότι συναπόφαση σημαίνει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο νομοθετικά όργανα και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμφωνήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα διευκολύνει με όλες τις δυνάμεις τη συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι, αφορά αυτό που είπε η κυρία Λόχμπιλ, ότι δεν υπάρχει ακόμα έγγραφο για την εισηγητή ε, και ότι θα να συζητήσει περισσότερο το περιεχόμενο της πρότασής μας στο πεδίο εφαρμογή με χαρά μου να κάνω αυτή τη συζήτηση με την κυρία Λόχμπιλ. Θα ήθελα απλώ να διαβεβαιώσω την Επιτροπή σας ότι στην πρότασή μας έχουμε βάλει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος. Συμφωνούμε για το ποιο είναι το πρόβλημα, συμφωνούμε για το ποια προγράμματα θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε με αυτό το μέσο. Εμείς έχουμε διατυπώσει τα πράγματα έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε <clears throat> να ε, επιτελέσουμε το έργο μας. Πάντως είμαι ανοιχτό ε, και μπορώ κάλλιστα να έχω μια διμερή επαφή με την κυρία Λόχμπιλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, αδίδω το λόγο στην κυρία Βαρβάρα Λόχμπιλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη που δεν έχω έγγραφο, αλλά ήταν δύσκολο. Όποτε προκύψει, όποτε το έχω, θα σας το προωθήσω, θα σας το διαβιβάσω. Και βεβαίως ε, σημείωσα ότι θα πρέπει να έχουμε συζήτηση με το Συμβούλιο για να διερευνήσουμε τις διάφορες νομικές απόψεις που υπάρχουν επί του θέματος. Αυτά στο παρόν στάδιο. Προσδοκώ στην στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους και εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και θα επιστρέψουμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ με ένα έγγραφο και ελπίζω να λάβω μέχρι τότε και μια σαφή αποκρισταλωμένη γραπτή θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και η συνθήκη της Λισαβόνας που θα έχει κατά πάσα πιθανότητα και ελπίδα τεθεί ενισχύ. Άρα συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση σας κυρία Λόχ Μπίλερ και αυτό προτείνω να εγκρίνει και η Επιτροπή μας. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την κυρία Μπράτνερ. Είναι καθοδόν. Καταφθάνει ο νουπο έπρεπε να υπάγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου έλαβαν χώρα κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, πέντε λεπτών υπομονή ζητώ για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεώς μας. Μην απομακρυνθείτε λοιπόν σας παρακαλώ, μην απομακρυνθείτε πολύ.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 Please. Let's move on. Παρακαλώ, να συνεχίσουμε. Όλοι. Λοιπόν, Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ζητήσω Μπραντνερ, την εισηγήτρια, να λάβει το λόγο και να μας πει αν υπάρχει κανένα θέμα για την ψηφοφορία. Καλημέρα. Guten Με συγχωρείτε γιατί καθυστέρησα. Στο αεροδρόμιο έγινε η καθυστέρηση γιατί ερχόμουν από τη Γερμανία και στη, εχθές όπως ξέρετε είχαμε τους εορτασμούς και αυτό καθυστέρησε τα πάντα. Λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πέντε λεπτά μόλις πριν λάβαμε το κείμενο της Κομισιόν όπου αναφέρεται η ανάγκη να περάσει η χρηματοδότηση από το 5% στο 10%. Και επίσης κάνει μια περιγραφή του στόχου της αύξησης αυτής. Επομένως εγώ που δέχομαι την πρόταση αυτή αποσύρω την τροπολογία μου όπου ζητούσα ακριβώς αυτή την αύξηση. Δεν χρειάζεται πλέον. Την είχε απορρίψει η Επιτροπή στην αρχή αλλά τώρα τη δέχεται και είπε ότι θα διανύμει και το καινούργιο κείμενο. Λοιπόν, ίσως ε, όσοι, όσοι όντως θέλουν το κείμενο να σηκώσουν το χέρι τους γιατί δεν έχω και τόσα πολλά αντίγραφα. Ναι, αλλά η, στο ΝΤΕΒΕ έχει κυκλοφορήσει. κυκλοφορήσει. Αναφέρομαι στο στρατηγικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, κυκλοφο... που διανύμεται τώρα. Ε, έφτασε ευτυχώς εν ε, για να αποσύρουμε την τροπολογία και αυτό είναι καλό και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έδωσε αυτό το έγγραφο είναι ένα καλό δείγμα συνεργασίας και ευχαριστώ, με τους, ευχαριστώ τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία. Ακούσαμε ότι η Ντεβε έχει ε, ε, υιοθετήσει μία τροπολογία η οποία μου λέτε ότι έχει κυκλοφορήσει και εμείς ε, θα θέλαμε να το τροπολογήσουμε γιατί μόνο 10% τώρα α, αναφέρεται στην ειρηνική συνεργασία και ε, μετά λέγεται ότι ε, γίνεται αναφορά στους ε, συνεργαζόμενους και θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στους εσωτερικούς πόρους. Γι' αυτό και θα ήθελα να προτείνω την εξής φράση. αρκεί η αύξηση να συνάδει με την αναθεώρηση της συνεργασίας και των εσωτερικών πόρων. Επαναλαμβάνω, αρκεί η αύξηση να συνάδει με ε, την ε, ε, τους εσωτερικούς πόρους και την αναθεώρηση της συνεργασίας. Ωραία. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Και εμείς θα θέλαμε να δηλώσουμε την ικανοποίησή μας λόγω του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέδωσε αυτή τη στρατηγική έκθεση την οποία είχαμε ζητήσει, την οποία είχε ζητήσει και η συγγήτρια και συμφωνούμε και με την προφορική τροπολογία που θα υποβάλει η συγγήτρια έναντι της τροπολογίας όπου εγκρίθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κέλαμ. Ε, εν ονόματι του ΕΛΚ πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μας διότι η συγγήτρια συνεφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αυξήσουμε το φάκελο χρηματοδότησης στο 10% ε, διότι δεν χρειάζεται να δένουμε τα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πρέπει να επεμβαίνει σε ορισμένες καταστάσεις. Συμφωνούμε με την εξήγηση ε, με την εξήγηση που παρουσίασε η κυρία Μπραντάουερ και χαίρομαι ιδιαίτερος που θα προχωρήσουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ρωτώ τους ε, συναδέλφους εάν ε, θέλετε να βάλετε την κάρτα σας ε, το, στη θέση της για να ψηφίσουμε. Αλλά η κυρία Λούνα Τσεκ θέλει να πει ότι εντωμεταξύ περιμένοντας την, την κάρτα θα ψηφίζω διαχειρός ε, και ε, είναι λόγω των εορτασμών στη Γερμανία. Ε. Εντάξει, δείξτε μας ποια είναι η θέση σας. Έχουμε την πρώτη, την πρώτη ψηφορία για την τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 3 και η προφορική 2 αποσύρονται. Τώρα έχουμε την ΤΕΒΕ 1 με την προφορική τροπολογία η οποία ε, υπερψηφίστηκε πριν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι ακόμη. Ωραία. Πρώτα οι κυρίες. Είμαι αδύναμος από αυτή την άποψη. Λίγη ψηφοφορία. Ψήφισαν 45 υπέρ και τρεις κατά και καμία αποχή. Συγχαίρω λοιπόν την εισηγήτρια και λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο ένα λεπτό να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες για την εξαιρετική συνεργασία. Προσβλέπω εις <clears throat> την συνέχιση της συνεργασίας στα επόμενα έτη. Ήταν όχι απλώς καλή, ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ.